υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Ο πρώτος που θα λάβει τον λόγο από τους συντάκτες ε, θα είναι η κυρία Χέντι Χάουταλα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά θα έπρεπε να ανάψουμε κεράκια τώρα και δεδομένων των δολοφονιών, της δολοφονίας ε, σε σχέση με την Τσετσένα ε, ε, υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον Άλεξ της Ζιμπραήλοβ ε, και την κυρία Σανταλάιεβα και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις Όλοι αυτά τα άτομα αξίζουν της υποστήριξής μας σίγουρα και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα και όταν βρισκόντουσαν εν ζωή Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εκφράσουμε την θλίψη μας και να πούμε ότι είναι ανησυχητικό, ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο το ότι δεν κατάφεραν οι ρωσικές αρχές να προβούν στην διευκρίνηση αυτών των περιστάσεων και γεγονότων αυτών των δολοφονιών και να προσαθούν στα δικαστήρια υπεύθυνοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απευθύνει διάφορα διαβήματα και επιστολές ε, στις ρωσικές αρχές, αλλά αυτά δεν υπάρχουν. Πρέπει να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε, να δούμε πώς μπορούμε να καταφέρουμε στη Ρωσία να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου και να είναι σεβαστή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει πολύ σοβαρότερα να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα όταν θα προβούμε σε νέε ε, συζητήσεις με τους Ρώσου ως εταίρο για μια νέα συμφωνία που θα διέπει τι σχέσει μας. Πρέπει να προβληματιστούμε να δούμε πώς καλύτερα από ότι στο παρελθόν μπορούν να προστατεύονται οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Πρέπει να δούμε αν μπορούμε να προσφέρουμε πραγματικά η προστασία σε άτομα που απειλούνται. Αν ταχύτατα μπορούν να υποβάλουν κάποιες προσφορές ε, σε αυτά τα άτομα ή ε, ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορούν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία αυτά τα άτομα και να προστατευτούν αλλού. Είναι σημαντικό στην Ευρωβουλή να υπάρξει ένα κέντρο όπου θα διαχέονται πληροφορίες και θα ενημερώνονται οι πολίτες σε σχέση με την κατάσταση των ανθρώπων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ρωσία. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Η Παλιτικόσκα είχε πει εν ζωή ότι η Δύση μπορεί πάρα πολλά να κάνει, αλλά πράττει πολύ λίγα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Χάουταλα. Επόμενο αγορητή, η κυρία Ντεκέζερ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ε, να ξεπίσω το λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου ε, για να παρουσιάσω τη θέση της ομάδας μου που ε, δεν συμφώνησε με το κοινό ψήφισμα και προτείνει ένα δικό, του, ένα δικό της ψήφισμα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι συμφωνούμε απόλυτα με το κοινό ψήφισμα όσον αφορά την Ναταλία Εσμυρινοβά, την ε, Ζαντούλιεβα ε, και τον Αλίκ Ζαμπράιλοφ. Πρέπει να σας πω ότι ε, αισθανθήκαμε φρίκη απέναντι σε αυτές τις ε, νέες δολοφονίες που είναι ε, ορισμένες ακόμα δολοφονίες ε, αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Τζετσενία. Στο ψήφισμά μας ζητήσαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ζητάμε το ίδιο ακριβώς πράγμα με το κοινό ψήφισμα. Δηλαδή καταδικάζουμε την επίθεση, ζητάμε να γίνει έρευνα, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των, ε, και των αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί που διαφορά είναι στο γεγονός ότι διευρύνεται ε, η αναφορά σε όλους τους, αγωνιστέ τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην κατάσταση στον Βόρειο Κάφκασο. Ε, γιατί νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει αλλού. Για παράδειγμα, στο ψήφισμα το οποίο θα προηγηθεί τη Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ρωσίας και θέλουμε αυτό το θέμα των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η περάσπισή του να ε, είναι μέρο του ψηφίσματο αλλά και να συνοδεύσει όλε τι διαπραγματεύσει με τη Ρωσία. Το διευκρινίζω λοιπόν. Εδώ αναφερόμαστε. Ε, το, για μα το πρόβλημα είναι πρόβλημα διαγράμματο και τόπου. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πολιτικό τρόπο. Και όχι μόνο εδώ στα κατεπήγοντα. Υπό αυτή την έννοια προτιμάμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Αλλά φυσικά, επί της ουσίας, συμφωνούμε απόλυτα με τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ρενάτε Βέμπερ στη συνέχεια παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω κάποια γεγονότα. Εφέτος μόνο τον Ιανουάριο ο Στανισλάβ Μαρκελόφ, ο συνήγορο υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εκπροσωπούσε την δολοφονηθήσα Παλιτκόφσκαγια, κατά μεσήμερο δολοφονήθηκε και η Αναστασία Βαρβούροβα, μια δημοσιογράφος που προσπάθησε να τον, να τον προστατεύσει και εκείνη πυροβολήθηκε. Τον Ιούλιο η Νατάλια Ισμέροβα, μια πολύ γνωστή υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βρέθηκε στην Ιγκουσετία μετά την απαγωγή της στην γειτονική Τσετσενία, βρέθηκε νεκρή εκεί. Στην συνέχεια, κάποιους μήνες μετά, ένας άλλος ακτιβιστής, η κυρία Σανταλάγεβα, απήχθη και δολοφονήθηκε και αυτή τον Αύγουστο δημοσιογράφος Κρυβιλόφ βρέθηκε νεκρός μόλις είχε εγκαταλείψει το σπίτι του. Έξι δημοσιογράφοι, όλοι εξέχουσες προσωπικότητες δολοφονήθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτές οι, αυτοί οι αλυσίδα δολοφονιών δείχνει ότι έχουν επιδεινωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και γίνεται προσπάθεια να θυμωθούν οι ανεξάρτητες φινές και αντιμετωπίζουν διωγμούς ε, όσοι προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και στο Βόρειο Κάυκασο δεν μπορούν να αγνοηθούν πλέον. Δεν μπορούμε να αμελούμε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και να θεωρούμε ότι με τις φιλοδοξίες υπερδύναμης η Ρωσία με μία από τις πιο αναπτυγμένες υπηρεσίες πληροφοριών παγκόσμια δεν είναι σε θέση να, προσαγάγει, να προσάξει στα δικαστήρια τους υπεύθυνου αυτών των περιπτώσεων. Πρέπει να δούμε ότι η ατιμορρησία όσον αφορά τις δολοφονίες αυτών των υπέρμαχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συνεισφέρει στην αύξηση της ε, βίας ακόμα περισσότερο. Οι ρωσικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν την σωματική προστασία αυτών των υπέρμαχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία κινήσεων του σύμφωνα με τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ισχύει από πλευρά ΟΗΕ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία. Στη συνέχεια ο κύριος Μπέρν Πόσερτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε ο προηγούμενος πρεσβή, πρεσβύτερος πρόεδρος στην Ευρωβουλή, όθων των Αψβούργων, ρωτήθηκε αν δεν εκφράζει την θλίψη του για το ότι δεν είναι αυτοκράτορ των Ευρωβουλευτών. Είπε όχι, δεν, είμαι, ε, δεν θλίβομαι γι' αυτό γιατί θα έπρεπε αν ήμουν αυτοκράτορας να αποκαλώ τον κάθε γάιδαρο εξοχότατε, ενώ τώρα μπορώ τον κάθε γάιδαρο να τον αποκαλώ γάιδαρο. Δεν πρέπει να είμαστε διπλωματικό σώμα, δεν είμαστε διπλωματικό σώμα, είμαστε ένα πολιτικό κοινοβουλευτικό σώμα και μπορούμε να λέμε απροκάλυπτα και στα ίσια ξεκάθαρα την αλήθεια. Υπάρχει ένα, μια παροιμία που λέει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και ευχαριστώ για την συνάδελφο, την συνάδελφο Βέμπερ που το εξέφρασε με αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι δολοφονίες, αυτά τα συμβάντα στον Κάφκασο δεν είναι τυχαία γεγονότα, ούτε είναι πράξεις κάποιων σκοτεινών δυνάμεων. Από την ανάληψη του αξιώματος που ε, κατέχει ο κύριος Πούτιν και από την έναρξη του προβλήματος της Τσετσενίας με τα, τους, τα, τις μυστηριώδεις εκρήξεις στη Μόσχα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ένα αιματηρό, ένα ματωμένο ίχνος που πάντα δείχνει τον δρόμο στην Τσετσενία και πλήττουν αυτές οι δολοφονίες αθώους, άμαχους και καμιά φορά υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που τους γνωρίζουμε λόγω της δράσης τους ε, και που ε, κατέβαλαν προσπάθειες ε, όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τσετσενία αλλά για μια δημοκρατική Ρωσία και την κατανόηση μεταξύ των λαών Τσετσενίας και Ρωσίας και για την ειρήνη στον Κάφκασο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα θύματα. Αυτοί ο ένας μετά τον άλλο δολοφονούνται και γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι, όπως από πλευράς ε, κατεπήγοντος θα γελιοποιούμεθα αν η κυρία η οποία μας, ε, ε, την, οποία βραβεύσαμε που ήρθε εδώ αν συνεχίζονται αυτές οι δολοφονίες και εμείς αναβάλουμε αυτή την υπόθεση για ιστερότερη συζήτηση στην Ρωσία βλέπουν πάρα πολύ καλά και προσέχουν αν είμαστε σε θέση άμεσα να αντιδράσουμε και πρέπει άμεσα να αντιδράσουμε και να πούμε φτάνει πια με αυτές τις δολοφονίες, φτάνει πια με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία για την Τσετσενία, ελευθερία για τη Ρωσία, αλλά να τερματιστούν οι συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτών των δολοφονιών <clears throat> μυστηριώδη πλαίσια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια ο κύριος Τόμασα Φορέρ. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα μια φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάμε για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Είναι ένα θέμα που επανέρχεται διαρκώς. Μιλάμε για τα βασανιστήρια και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν ε, ε, απειλές και δολοφονία πλέον στη Ρωσία. Οι έρευνες δεν καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα Μιλάμε για απαντελή έλλειψη αποτελεσματικότητα. Ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να είναι το στοιχείο κλειδί στι σχέσει μα με τη Ρωσία. Έχουμε υποχρέωση να απαιτήσουμε από τη Ρωσία να ξεκινήσει ε, διαδικασία ανακρίσεων ερευνών και να οδηγήσει του υπεύθυνου στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενο ομιλητή, η κυρία Κορνέλια Έρνστ, για δύο λεπτά. Μάλιστα κυρίε και κύριοι, επιτρέψτε μου ως νέα Ευρωβουλευτή να μπορέσω να διαπιστώσω ότι σε κάποια νομικά θέματα και για τη δική μου ομάδα την γερμανική αριστερά Deutsche Linke διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και ότι κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να καταδικάζεται ανεξάρτητα από το που συμβαίνει και ποιοι την ε, προκάλεσαν. Δεν έχει τίποτα κάτι τέτοιο με την ανάμειξη σε εσωτερικές υποθέσεις ενός άλλου κράτους. Πραγματικά ανησυχώ και εδώ και πολλά χρόνια και εξοργίζομαι ότι δολοφονούνται ε, υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασχολήθηκαν με την κατάσταση στην Τσετσενία. Νατάλια Εστεμίροβα, Κόρνιλοφ, Σανταλάγεβα Αυτά είναι παραδείγματα για το τι συμβαίνει πρέπει να μας συγκλονίζουν και πραγματικά κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να απασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση και θα ήθελα να πω ότι με ανησυχεί ιδιαίτερα ότι δεν, δεν εξηχνιάζονται τέτοιες δολοφονίες, ούτε της Άννας Παλιτκόφσκαγια. Και τώρα όταν ξαναρχίζει αυτή η δίκη για τη δολοφονία της, ελπίζω πράγματι ειλικρινά ότι θα προσαχθούν στα δικαστήρια οι υπεύθυνοι, διότι διαφορετικά με ατιμορρησία νέες τέτοιες δολοφονίες επαπειλούνται. Αυτό που αναμένουμε είναι απλό. Θέλουμε άμεσα κάθετα να ζητήσουμε να εξηχνιαστούν αυτοί οι φόνοι. Και μάλιστα χωρίς κανένα έλεος. Άτεγκτα πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να αναπεριμένει κανείς. Ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να εγγραφεί στα ίδια μας τα λάβαρα. Δεν είναι δυνατόν η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να οδηγεί κάποιους ανθρώπους σε θάνατο και σε δολοφονίες και πρέπει η κορυφή η, με τη Ρωσία να απασχοληθεί με αυτά τα θέματα άμεσα, όχι κάποτε αλλά άμεσα και με την πρώτη ευκαιρία. Θέλουμε η αντιμετώπιση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων να γίνει με αυτόν τον τρόπο και δεν θέλουμε να εξετάζεται το θέμα στο περιθώριο. Και μόνο τότε όσον αφορά το εμπόριο και τις ε, οικονομικές σχέσεις ε, δεν πρέπει να εξετάζουμε τέτοια θέματα ως δευτερεύοντα αλλά ως πρωτεύοντα. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε μια χώρα με τόσο πληθυσμό κάποιοι πεθαίνουν τυχαία σαν θύματα της ε, συνήθους εγκληματικότητας αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι επίθεση της ε, Ρωσίας κατά της Πολωνίας ε, τεράστιος αριθμός Πολωνών πολιτών θανατώθηκε τη στιγμή εκείνη αυτά τα γεγονότα θεωρήθηκαν σαν κάτι το κοινότυπο όπως και η δολοφονία των, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αύξηση αυτών των δολοφονιών μας δείχνει ότι αυτό, η αντίληψή μας για αυτό το φαινόμενο αυτό είναι τελείως εσφαλμένη. Μιλάμε για το συστηματικός χαρακτήρας αυτών των δολοφονιών δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη Ρωσία με αποτέλεσμα να είναι αυτές οι δολοφονίες, αυτά τα εγκλήματα τόσο συχνά. Η επέκταση του φαινομένου είναι αποτέλεσμα της βαθιάς ηθικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Το ψήφισμά μα είναι ισορροπημένο και θα μα επιτρέψει να κάνουμε ένα βήμα προ την επίλυση αυτού του προβλήματο. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριο Παλέκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. και η δική μου ομάδα προβληματίζεται με αυτά που συμβαίνουν στη Ρωσία. Η Νατάλια Στεμίρεβα, η Πολιτόσκαγια, η Μαλάιωβα και όλοι και πολλοί άλλοι δολοφονήθηκαν. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, να καταδικάζουμε τους υπεύθυνους για αυτές τις δολοφονίες γιατί να υπάρχει αυτό το κλίμα ατιμορρησίας σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας. Ο πρόεδρος ο Ρώσος, ο κ. Μετβέντεφ, υποσχέθηκε ότι θα αναζητήσει και θα βρει εκείνους που ευθύνονται για αυτές τις δολοφονίες. Μίλησε με περισσότερη έμφαση σε σχέση με τον προηγούμενο πρόεδρο, αλλά έμεινε στα λόγια. Ο χρόνος θα δείξει αν θα τηρήσει την υπόσχεσή του και αν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε τις ε, πράξεις της Ρωσίας στο Νότιο Κάφκασο οι σοσιαλιστές και δημοκρατικοί αποφάσισαν να προωθήσουν το δικό τους έγγραφο. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία θα μπορούσε να βελτιωθεί εάν γίνουν διαβουλεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις παράλληλα με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ε, ρωσικούς κρατικούς, ε, κρατικούς φορείς είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό το οποίο, στο οποίο πρέπει να παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, η κυρία Αντρικένα. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή ε, και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι δολοφονίες των ε, προεσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία είναι πάρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή όπου διαρκώ φτάνουν στα αυτιά μας δολοφονίες ε, ε, αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Σαντουλάγεβα, ο Τζαμπράιλοφ και άλλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αγνοεί αυτή, αυτή την κτηνώδη συμπεριφορά ε, και αυτές ε, τις δολοφονίες των προσφυστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε κάθε μας επαφή λοιπόν με τη Ρωσία πρέπει να τους υπενθυμίζουμε ότι οι έρευνες παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και ε, σε τελευταία ανάλυση οι ένοχοι δεν προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό είναι ο κανόνας, αλλά αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ιδιαίτερα στην περίπτωση, όταν μιλάμε για την Τσετσενία, όπου πραγματικά η εγκληματικότητα είναι πάρα πολύ υψηλή. Πάντα πρέπει να υπερασπίζουμε τι βασικέ μα αρχέ ανθρώπινη αξιοπρέπεια ε, και του δικαιώματο στη ζωή. Δεν υπάρχουν άλλε αξίε που να είναι, πιο, ε, που να είναι ανώτερε από τι αξίε αυτέ. Πρέπει λοιπόν να ε, φροντίσουμε να, και να πιέσουμε έτσι ώστε να συνεχίσουν οι έρευνε και να προσαχθούν οι ύποπτε στη δικαιοσύνη. Σα ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή, ο κύριο Κέλλαμ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία έχει αλλάξει ε, προς το χειρότερο. Ε, πρέπει λοιπόν να ε, πιέσουμε τι αρχέ τη Ρωσία ώστε να, καταβάλουμε, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διορθωθεί η κατάσταση. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό που λείπει είναι η βούληση. Μπορούν να γίνουν πολλά όταν όμως το Κρεμλίνο θα ασκήσει αποφασιστικό ε, έλεγχο ε, στις κρατικές δομές και στη δικαστική εξουσία. Ακριβώς επειδή η δικαστική εξουσία, ε, το δικαστικό σύστημα της Ρωσίας δεν μπορεί να υπερασπίσει τους ανθρώπους αυτούς, καταλαβαίνετε, γι' αυτό το λόγο η ευθύνη του καθεστώτος είναι μεγάλη. Πρέπει λοιπόν να, το μήνυμα να είναι σαφές. Όσο το, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να αφήνει αυτή την κατάσταση ε, και παραμένει μόνο στις δηλώσεις καλών προθέσεων, δεν μπορούν να βελτιωθούν οι οικονομικές μας σχέσεις. Ε, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Ρωσίας πρέπει να καταλάβουν ότι, ε, ότι η, Ευρωπαϊκή Ένωση άντισε τα συμπεράσματα που έπρεπε από, το κτηνόδι, από την κτηνόδη δολοφονία της Πολιτόφσκα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σόνικ έχει το λόγο στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Είναι μια συμβολική σημασία σήμερα όταν κάνουμε λόγο για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν από 7 χρόνια ο Ερυθρός στρατός, από, πριν από ε, το 1939 ε, ξεκίνησε η κατοχή των σταλινικών δυνάμεων και των χιτλερικών δυνάμεων του πολωνικού εδάφους. Υπήρξαν ε, χιλιάδες δολοφονίες και χιλιάδες Πολωνοί αξιωματικοί δολοφονήθηκαν στο Κατίν και βλέπουμε ότι η ημέρα αυτή θα είναι μια ημέρα ντροπή για τη Ρωσία. Σήμερα δεν μπορεί η Ρωσία να αντιμετωπίσει το ίδιο της στο παρελθόν και μέχρι σήμερα η Μόσχα δεν άνοιξε τα αρχεία της και δεν έδωσε καμιά πληροφορία για τις δολοφονίες του Κατίν. Στην ιστορία κάθε κράτους, κάθε χώρας υπάρχουν τρομερές στιγμές. Όμως θα πρέπει να έχει το θάρρος μια χώρα να αντιμετωπίσει το παρελθόν της. Όπως η Γερμανία για παράδειγμα. Μόνο με αυτό το θάρρος μπορεί να πάψει το παρελθόν, να διώκει το παρόν, να διώκει το παρελθόν της Ρωσίας στη σημερινή Ρωσία. Μόνο αν κοιτάξουν κατάματα το παρελθόν τους οι Ρώσοι και μόνο έτσι θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τη σταλινική κληρονομιά και θα πάψουν να πολεμούν εναντίον των ιδίων των πολιτών τους, πολιτών που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. <clears throat> Αυτοί που δολοφονήθηκαν είναι θύματα τα οποία θα τα θυμόμαστε πάντα. Δόξα σε αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταβάρες παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Η δολοφονία που αναφέρθηκε παρακολουθήθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση από όλους μας μόλις μάθαμε ότι είχε απαχθεί και ακούσαμε για αυτό το έγκλημα και μετά βρέθηκε δολοφονημένη. Είναι κάτι που δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο κανέναν οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο. Και η, ε, όπως αναφέρθηκε πιο πριν πραγματικά θεωρώ ότι η αριστερά πρέπει να υπερασπίζεται τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπουδήποτε και αν βρίσκονται και παντού να τους, υπερασπιζόμαστε. Οι επιπτώσεις αυτών των επιθέσεων κατά των υπερμάχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, οι επιθέσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Λειτουργούν ως μέτρο εκφοβισμού και σίγουρα είναι τραυματι... πράξεις που τραυματίζουν τους ε, ανθρώπους ε, και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια πρώτη φάση μια επίθεσης που επιδεινώνει μετά στη συνέχεια όλη την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέρα από τα δικαιώματα των ιδίων των ακτιβιστών. Οι επιπτώσεις αυτών των δολοφιών αιώνα ε, είναι πραγματικά πρόβλεπτες και είναι πολύ ομές. Χωρίς μια δικαστική εξυχνίαση αυτών των περιπτώσεων, χωρίς εγγύσει ότι η ασφάλεια των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα διασφαλίζεται δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια ομαλή εξέλιξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Γι' αυτό θα υπερψηφίσουμε αυτή την πρόταση ψηφίσματο. Και στη συνέχεια απευθύνουμε έκκληση στι αρχέ τη Ρωσία να προστατεύουν του υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ προέρχομαι από την Πορτογαλία, από το άκρο της Δυτικής Ευρώπης, αντιδιαμετρικά αντίθετο σε σχέση με τη Ρωσία γεωγραφικά. Και πιστεύω ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας έχουν τεράστια σημασία και η Ευρώπη οφείλει πολλά στη Ρωσία. Το πρώτο πράγμα το οποίο οφείλει είναι, οφείλεται είναι αποσαφήνιση των πλαισίων αυτών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης και των πολιτών της Ρωσίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία του Catch the Eye. Ο πρώτος ομιλητής, ομιλητής είναι η κυρία Κόρχουλα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, και πάλι. Είναι καλό να μπορώ να ομιλώ στην μητρική μου γλώσσα θα ήθελα να αντιδράσω στην δική σας παρέμβαση, συνάδελφε. Είναι σαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι παραβιάσεις τους να ήταν ένα πρόβλημα το οποίο αφορά μόνο την αριστερά. Όχι. Είναι κοινό ε, μέλημα και ε, όλοι ενδιαφερόμαστε σε αυτά, για αυτά. Συζητούμε εδώ στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, ενώ πάμπολοι έχουν φύγει ήδη για να επιστρέψουν στην ε, χώρα τους και η Ολομέλεια είναι άδεια. Είναι όμως σημαντικότατα θέμα θέματα αυτά. Ήμουν στο παρελθόν μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΑΦΕΤ και όταν, συνεδρίαζε, όταν δημιουργήθηκε, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχα και εκεί συνεργάστηκα και πολλοί από εμά έλεγαν στην υποεπιτροπή γιατί τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξετάζονται σε αυτό το πλαίσιο, ενώ θα έπρεπε να εξετάζονται στο πλαίσιο της υποεπιτροπής, έλεγαν πολλοί. Δεν αληθεύει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει αυτό να γίνεται. Σαν να είναι δηλαδή η υποεπιτροπή μας ένα γκέτο, όπου μόνο εκεί μπορούν να μετατεθούν τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για να επιληθούν αυτά τα θέματα. Στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω στον κύριο Πόσελτ. αυτά που μας είπε η κυρία Ντεκάιζερ για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι κάτι που μπορεί οποιοδήποτε να αμφισβητήσει ήταν πάντοτε κάποια που αναλάμβανε πλήρως τις ευθύνες της. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτά που είπε οι σοσιαλιστές ε, και τις θέσεις των σοσιαλιστών δημοκρατικών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προασπίζαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν εσείς κύριε Πόσελ προσπαθούσατε να κάνετε ότι δεν γνωρίζατε αυτά που συνέβαιναν στο Ιράκ ή στο Γκουαντάναμο. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία πρόκειται για ένα σοβαρότατο πρόβλημα και το σχέδιο ψηφίσματός μας είναι σαφές. Ωστόσο πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει τα θέματα ένα προς ένα και να μην υποβάλει κατάλογο αιτημάτων ε, απλά στη Ρωσία χωρίς να περιμένει κανένα αποτέλεσμα. Μια αντιπροσωπεία σοσιαλιστών και δημοκρατικών θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα τη Μόσχα και θα θέσουμε το ερώτημα με πολύ σαφή και συγκεκριμένο τρόπο ας μην εκμεταλλευόμαστε καταστάσεις όπως τη σημερινή για να ετοιμάσουμε απλώς έναν κατάλογο προβλημάτων που δεν θα συζητηθούν ποτέ με τις ρωσικές αρχές. Ας εστιαστούμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ανησυχία μου για τα συμβάντα τα οποία τον Ιούνιο συνέβησαν στην Ομοσπονδία της Ρωσίας. Συγκλονιζόμαστε από τις δολοφονίες ε, της Νατάλια Εστεμίροβα και Κουλάγιν που ήταν υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα λοιπόν ώστε να καταφέρουμε οι υπεύθυνοι να ε, βρεθούν και να προσαχθούν στα δικαστήρια. Όσον αφορά την παραβίαση διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων, συνέβη και αυτό σε σχέση με την σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και της Γεωργίας είναι λοιπόν αναγκαίο για όλους αυτούς τους λόγους η κυβέρνηση της Ρωσίας να τοποθετηθεί κάθετα επ' αυτών και να πει ότι καταδικάζει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν θα την ανέχεται πλέον. Κύριε Στάνοκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η ατιμορρησία που σημαίνεται στη Ρωσία όσον αφορά τα όσα συμβαίνουν κατά των ε, υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διώκονται δημοσιογράφοι, εθνικές μειονότητες ε, υφίστανται κάθε δίωξη και όλα αυτά συνεχίζονται. Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καλύτερη περίπτωση περιθωριοποιούνται, στην χειρότερη περίπτωση φημώνονται ή δολοφονούνται. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Ρωσία και επανειλημμένα βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα γεγονότα παραμένουν ατιμόρυτοι. Είναι συνηθισμένη η Ρωσία στο να λαμβάνει απλά υπόψη η Ευρώπη αυτά τα γεγονότα και να μην αντιδρά όπως και για την εισβολή στη Γεωργία των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων ε, πέρσι και δεν έγινε τίποτα. Και ενδιαφέρονται βέβαια οι Ευρωπαίοι να έχουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Όμως αυτό δεν μπορεί να μας παρακολύσει από το να θίξουμε αυτά τα θέματα και να είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών της Ευρώπης, της, της Ρωσίας που πρέπει να διασφαλίζεται ακριβώς αυτή η πτυχή. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Μόρβαϊ παρακαλώ ένα λεπτό. Ε, σας ευχαριστώ. Για 25 χρόνια είμαι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως δικηγόρος και γι' αυτό πρέπει να πω ότι ομιλώ και με συγκλονίζει και εκφράζω τα συναισθήματά μου για τους συναδέφους για αυτό το ε, αγαθό, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκφράζω πραγματικά την θλίψη μου για την απώλεια των οικείων τους στις οικογένειές τους. Τι πρέπει να γίνει. Νομίζω πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει δικαστική διερεύνηση και να υπάρξει αποσαφήνιση αυτών των γεγονότων από τις κρατικές αρχές χωρίς καθυστέρηση. Και ελπίζω ειλικρινά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θεμητοποιείται και νομιμοποιείται να κάνει κάτι τέτοιο. Όμως φοβούμαι ότι κάτι τέτοιο δυστυχώς μπορεί να μην συμβεί. Και γιατί. Διότι απλά και μόνο έχουμε αιτήματα έναντι άλλων χωρών. Αλλά αν κάτι συμβαίνει μέσα στο ένα ίδιο το ε, κράτο μα, όπω στη δική μα χώρα, για παράδειγμα στην Ουγγαρία, παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κύριο Παλ Σμιτ, ο αντιπρόεδρο, γνωρίζει φυσικά το τι τεκταίνεται και τι συμβαίνει. Διαδηλώσει που από δεκάδε χιλιάδε άτομα διοργανώθηκαν για να θυμηθούμε την Επανάσταση του 1956 στην Ουγγαρία και τι συνέβη. Συνέβησαν πράγματα τα οποία δεν διερευνήθηκαν δεν διερευνήθηκαν ακόμα από το κοινοβούλιο μας. Και εφόσον συνεχίζουμε μια τέτοια πορεία, έχουμε έναν αντιπρόεδρο σε μια υποεπιτροπή που ήταν μέρος ε, της, μέλος της κυβέρνησης που ήταν υπεύθυνη για τα όσα συνέβησαν και δεν θεμητοποιούμεθα για να εκφράζουμε απόψεις έναντι τρίτων χωρών για την προστασία των ε, διοκόμενων και για να αποσαφινιστούν ε, τα όσα έχουν συμβεί. Αυτό πρέπει να το δούμε σε σχέση και με την Ουγγαρία για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ χρησιμοποιείται περισσότερο χρόνο, χρησιμοποίησαμε περισσότερο χρόνο από ό,τι είχαμε υπόψη για αυτό το θέμα. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει κάθε ένας να έχει την ευκαιρία να εκφραστεί και ζητώ την κατανόησή σας. Ο κύριος Πρέντα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα καταρχάς να πω ότι με απογοήτευσε το γεγονός ότι όταν μιλούσαμε για την κρίση για το γά, του γάρακτος ήταν γεμάτη αίθουσα, ενώ τώρα που μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε 40 δεν είμαστε παρόντες. Κρίμα. Όχι ότι το γάλα δεν είναι σημαντικό ζήτημα, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, δεν είναι αμεληταία πολιτικά. Να πω επίσης ότι φέτος, όπως γνωρίζετε, πολλές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης γιορτάζουν τα 20 χρόνια της πτώσης του κομμουνισμού. Η ιδέα ότι τόσο κοντά σε μας μία δύναμη από την οποία γεννήθηκε ο κομμουνισμός δείχνει τέτοια διαφορία για τα εγκλήματα κατά των αγωνιστών για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι κάτι το απαράδεκτο. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να δηλώσουμε το ότι ο, η, ο ολοκληρωτισμός πρέπει να απομακρυνθεί άπαξ διαπαντός. Πρόεδρος, τελείωσε η... τελείωσαν οι αγορητέ και ζητώ από την κυρία Κούνεβα να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση για την κατάσταση των αγωνιστών για τα δικαιώματα του ανθρώπου στη Ρωσία είναι πολύ ισορροπημένη και σωστή. Ε, οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί στην δουλειά τους. Πολλοί πλήρωσαν με τη ζωή τους το, το, το τίμημα της ε, καταγγελίας της παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα ήθελα να αποτίσουμε τιμή σε όλους όσοι έδωσαν τη ζωή τους και σε όλους όσοι συνεχίζουν να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Πολλά Πολλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου έγιναν χώρα στο Βόρειο Κάφκασο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολλού από του ανθρώπου που είναι τέρημα στην εφαρμογή έργων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αθώοι πολίτες, προσωπικό της, ε, ε, του, νόμου και απλοί πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη μάχη αυτή. Η βία κατά των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν περιορίζεται μόνο στο Βόρειο Κάφκασο. Υπάρχουν αναφορές ότι δικηγόροι, αγωνιστές και ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι σε όλη την Ρωσική Ομοσπονδία αντιμετωπίζουν βία παρενόχληση και εκφοβισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να μιλά κατά των παραβιάσεων αυτό και να τονίζει ότι η Ρωσία πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι κρίσιμο η, η, ε- η βίαιη θάνατη αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τύχουν σωστή έρευνας και οι δράστες να αναζητηθούν και να τιμωρηθούν. Μόνο μέσω πραγματικής δίωξη των, θανάτων, των ε, δολοφονιών αυτών θα σταματήσει η ατιμορρησία και η βία. Ο πρόεδρος Μετβέντεφ μίλησε κατά του νομικού μηδενισμού όπως τον χαρακτήρισε που κυριαρχεί στη Ρωσία και πρέπει να υποστηρίξουμε στη Ρωσία στην, μετα... συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρεί πολύ σημαντική την ε, συζήτηση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διάλογο της με τη Ρωσία και καλωσορίζει την ανοιχτή θέση που έλαβε ο πρόεδρος Μεντβέντεφ στη συζήτηση με την Ένωση για τα θέματα αυτά. Η επόμενη Σύνοδος Κορυφή Ένωση Ρωσία είναι μια άλλη ευκαιρία για να συνεχιστούν οι συζητήσεις αυτές. Τούτο πρέπει να συμπληρώνεται από μια ανταλλαγή μεταξύ πυρογνωμόνων. Οι διαβουλεύσει Ένωση Ρωσία προσφέρουν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα αυτό και να να ζητήσουμε συνομιλητές συζητήσεων θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ασφάλεια των αγωνιστών για τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να είναι η πρώτη μας μέρημνα. Ζητούμε από τις ρωσικέ αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν τόσο να εξασφαλίσουν πως όσοι εργάζονται για να δοθεί, να εμφανιστεί φως στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή, μπορούν να το κάνουν χωρίς φόβο βίας ή εκφοβισμού. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Προχωρούμε τώρα στη συζήτηση πέντε σχεδίων ψηφίσματος για το Καζακστάν. Ιδιαίτερα δε την περίπτωση του Γευγένη Ζόφτης. Οι συντάκτες. Η κυρία Χάουτελα, δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω